Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a... Uh, Κυρίες και κύριοι, τρεις και μία. Ξεκινάμε. Σημείο 9 στην μερίσια διάταξη. Η στρατηγική της Ένωσης κατά της αποψήλωσης των δασών. έγγραφο 2019-352 της Κομισιόν που ετοίμασε η Επιτροπή και έχει μπει πλέον στην δημόσια διαβούλευση. Από ό,τι φαίνεται, από το 90 έως το 16, κάθε ώρα χάναμε δάσος μεγέθους 800 γηπέδων ποδοσφαίρου κάθε ώρα. Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει ζήτηση προφανώς, πρωτεσίλες, ξύλο, μεγάλες, ε, μεγάλη ζήτηση για ξύλο, το σόγια. Αλλά η αποψήλωση των δασών έχει συνέπειες. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μια σχετική στρατηγική. Βέβαια υπάρχουν κάποια ελλειπή μέτρα κατά της ε, ανέλεγκτης αποψήλωσης των δασών, το φλέκτ, αλλά από ό,τι φαίνεται μόνο η Ινδονησία προς το παρόν ξεκίνησε να εκδίδει αυτά, αυτές τις άδειες με την ειδική επισήμανση. Από την οπτική της Ένωσης θα χρειάζονται και άλλες ε, δράσεις. Έχουμε την Άστριτ Σούμαχερ από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος υπεύθυνη για την αποψήλωση του, των δασών και την συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση επίσης Περιβάλλοντος. Η Άστριτ πρώτα έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για την εισαγωγή. Το θέμα συζητείται βέβαια και σήμερα στην ε, Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα στην Νέα Υόρκη. Εγώ θα σας παρουσιάσω ένα κείμενο αντίστοιχο περίπου με αυτά που είχα πει στην Επιτροπή Envy. Προτείνω σε τρία μέρη να σας ενημερώσω για την ανακοίνωση, να πω δύο λόγια για το FLECT, ε, που είναι ένα υφιστάμενο εργαλείο, και η συνάδελφος από το Trade θα έρθει με κάποιες γενικότερες συζητήσεις για τη σχέση μεταξύ εμπορίου, εμπορικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και πώς αυτές οι δύο κατηγορίες πολιτικών μπορούν να συνυπάρξουν. Να σας δώσω το πλαίσιο. Μιλήσατε ήδη για τα 800 γήπεδα ποδοσφαίρου δάσους που χάνουμε κάθε ώρα. Τα δάση αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο και από την αποψήλωση και από την υποβάθμιση των δασών. Οι φωτιές του Αμαζονίου έδωσαν ε, πολιτικό μήνυμα, αλλά δεν ήταν οι μόνες φωτιές φέτος. Είχαμε τεράστιες πυρκαγιές στη Σιβηρία, σε μέρη της Αφρικής και στην Ινδία. 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους χάθηκαν από το 90 και μετά. Στην Ένωση η τάση είναι θετική. Τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε αύξηση της δασοκάλυψης. Τώρα, γιατί είναι σημαντικά και μας ανησυχούν όλα αυτά. Διότι τα δάση καλύπτουν 80% της βιοπικιλότητας, ε, της χερσαίας βιοπικιλότητας και έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία για το κλίμα. Η χρήση γης λόγω αποψήλωσης καλύπτει 12% της παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα. Η ανάληψη δράσης κατά της αποψήλωσης των δασών σημαίνει ανάληψη δράσης και κατά της αλλαγής του κλίματος. Ε, το 1 τέταρτο δε του πληθυσμού της γης εξαρτάται έμεσα ή άμεσα από το δάσος. Θα έχουμε λοιπόν ε, κρίσεις που είναι πολλών ειδών, φτώχειας, ε, κοινωνικού χαρακτήρα κλπ. Είναι σημαντικά να είναι σαφές λοιπόν τι οδηγεί την, στην υποβάθμιση του δάσους και την αποψήλωση των δασών. Πρέπει να πούμε ότι η αύξηση ζήτησης για τρόφιμα, ξύλα, ενέργεια και η αύξηση του πληθυσμού, ιδίως της μεσαίας τάξης ανά τον κόσμο, είναι ο κύριος λόγος. 20% της αποψήλωσης των ε, δασών αφορά ε, ισχύει λόγω της επέκτασης της γεωργίας. Δεν φταίει μόνο η γεωργία, αλλά υπάρχουν και ε, η αύξηση της ορυκτής παραγωγής κλπ. Υπάρχουν και ε, ενδογενείς λόγοι κλιματικού χαρακτήρα κυρίω, αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες και άρα χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για την εντόπιση των μέτρων, ε, για την εντόπιση του προβλήματος με πολλά συγκεκριμένα μέτρα. Συνολικά, τι κάνει η Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να λάβουμε δράση. 10% των προϊόντων της παραγωγής σχετίζονται με την αποψήλωση των δασών και την ένωση. Αυτό είναι σημαντικό και μας δίνει και εργαλεία να δουλέψουμε και ευθύνες όταν καταλάβουμε ιδίω ότι το μέρος του 10% στο συνολικό εμπόριο των ε, προϊόντων, των αγαθών, είναι σε ένα τρίτο ευρωπαϊκό. Σας είπα, ε, καουτσούκ, ξύλο κλπ. Επίσης, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία αυξάνουν τη ζήτησή τους σε προϊόντα που σχετίζονται με το δάσος, άρα η συμμετοχή της Ευρώπης θα περιοριστεί. Τώρα, το κείμενο της Επιτροπής που είχε υποβληθεί πριν τη σύνοδο του ΣΥΜΠΙΟΥ είχε τονίσει ότι η απώλεια των δασών δεν είναι πρόβλημα άλλων, είναι και δικό μας και πρέπει να είμαστε μέρος της λύσης. Όχι μόνοι μας, αλλά ως, είτε ως καθοδηγητές, είτε ως συνεργαζόμενοι για τη λύση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η πρόθεση της ανακοίνωσής μας είναι να δείξει τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Το κείμενο δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και έδειξε τι μπορεί να πώς μπορεί να συμβάλλει η Ευρώπη με άλλους στην αντιμετώπιση της αποψήλωσης των δασών. Ο στόχος μας ήταν ήδη από παλιότερα να μειώσουμε την αποψήλωση κατά 50% μέχρι το 2020, αύριο δηλαδή, και μια σειρά εργαλείων. Το light motive πίσω από αυτό είναι το partnership. Όχι δηλαδή μία δράση της Ένωσης μόνο, αλλά σε συνεργασία με άλλες χώρες, με άλλους καταναλωτές. Πέντε προτεραιότητες και 36 δράσεις ε, περιλάβαμε στην ανακοίνωση, αλλά σε ένα παράτημα υπάρχουν και συγκεκριμένα μέτρα για τις αρχές αλλά και για την κοινωνία των πολιτών. Οι πέντε προτεραιότητες πάω Οι πέντε προτεραιότητες υπάγονται σε πέντε τομείς. Ζήτηση, κατανάλωση, το, οι, οι, οι συνέπειες της κατανάλωσης, διεθνής συνεργασία, χρηματοδότηση και έρευνα ξεκινούμε εξετάζοντας την, τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ε, της Ένωσης, που είναι αυτό που έχει τη βασική ε, ευρωπαϊκή συμβολή. Πρέπει να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας πρώτα-πρώτα. Και αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε μια πλατφόρμα εμπλεκομένων, ούτως ώστε κάτι που προτείνουμε να λειτουργεί για όλους και να, ακούγουμε, να ακούγονται από όλους. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα πρώτα με εθελούσια συμμετοχή και κατόπιν, αυτό έχει γίνει και μέσα στο πλαίσιο του ΦΛΕΚΤ, και μετά θέλουμε να εξετάσουμε την επιπρόσθετη ζήτηση, αν χρειαστεί, με τους εμπλεκόμενους. Συνεργασία με τις χώρες παραγωγούς το πάω γρήγορα. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε μόνοι μας, χρειάζεται πολιτικό διάλογο, χρειάζεται να καθοδηγήσουμε την υποστήριξη και την χρηματοδότηση στην, στις χώρες παραγωγής, προστατεύοντας τα δάση και να προσπαθήσουμε να έχουμε μία σχετική βεβαιότητα ότι οι δράσει ανάπτυξη που χρηματοδοτούμε δεν θα οδηγήσουν το αντίθετο μάλλον σε ε, αποψήλωση. Διεθνή συνεργασία, αυτό είναι και δική σας αρμοδιότητα εδώ τη επιτροπή. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί, ιδίω ενθαρρύνοντας τη συνεκτική δράση με άλλες χώρες καταναλωτές ε, σε όλη την αλυσίδα ε, του προϊόντος. Άρα να αναλάβουμε δράση πολυμερός στο πλαίσιο του ΟΗΕ, τη Σύμβαση για την Βιοποικιλότητα, τη Γενική την Περιβαλλοντική Συνέλευση του, του ΟΗΕ, ό,τι θέλετε, για την αντιμετώπιση της αποψήλωσης και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που παρέχει η εμπορική πολιτική για το σκοπό αυτό. Επίσης πρέπει να ε, συζητήσουμε με τα κράτη την βιώσιμη χρηματοδότηση μέτρων κατά της αποψήλωσης και άλλα μέτρα, που είναι βιώ... άλλα μέτρα χρηματοδότησης που... και επενδύσεων που είναι ε, βιώσιμα και επιτρέπουν συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα. Έρευα και κοινωνία εντάχει. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και γι' αυτό θεωρούμε πολύ σημαντική δράση να υπάρξει ένα παρατηρητήριο της Ένωσης για την αποψήλωση του δάσους που θα μας βοηθήσει και εμάς και τις εμπλεκόμενες χώρες για την παρακολούθηση των εξελίξεων, των αλλαγών, των αιτιών και μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στην ενημέρωση για όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα της αποψήλωσης. Επόμενα βήματα. Μια μεγάλη διάσκεψη για τα δάση τον Ιανουάριο για να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό, δημιουργία μιας πλατφόρμας εμπλεκομένων, αξιολόγηση της, της επιπρόσθετης ζήτησης κυρίως ε, σαν θέμα προτεραιότητας και η δημιουργία του παρατηρητηρίου της Ένωσης, που είναι βάση για τα περισσότερα. Αυτό ήθελα να σας πω για την ανακοίνωση αυτή καθεαυτή. Να σας πω δύο λόγια αν έχω ένα λεπτό για το FLECT, Forest Law Enforcement Governments and Trade, ένα εργαλείο πολιτικής που υπάρχει από το 2003 ε, πριν ε, ο οικοτουρισμός γίνει φημίτες πάνω από κτήση γίνει της μόδας, είναι μια προσέγγιση που έχει στόχο την ανάπτυξη με περιβαλλοντική προστασία. Στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι να υπάρξει ένας κανονισμός για την ξυλία που αποκλείει την παράνομη ε, κοπή ξύλων, δημιουργεί εθελούσιες συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης, VPA, που επιτρέπει στις διμερίσεις εμπορικές συμφωνίες να εξάγουν προϊόντα, που επιτρέπει μέσω των διμερών συμφωνίων να εξάγονται προϊόντα με άδεια φλεκτ. Ακόμα πιο γρήγορα θα πάω εδώ, Πρόεδρε. Μία χώρα μόνο το έχουμε κάνει ακόμα, την Ινδονησία. Άλλες δύο, Γκάνα, Βιετνάμ, δουλεύουμε στενά προς την κατεύθυνση εκείνη για την αδειοδότηση FLECT. Άλλες χώρες, πολλές άλλες χώρες έχουν, ενδιαφέρονται. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι αν δόθηκαν και πόσες άδειες δόθηκαν, αλλά αν αυξήθηκε η ζήτηση για τέτοιες άδειες και αν τελικά το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Για την gracias. Thank you very much. Ευχαριστώ. Εμείς δεν θα ευθυγραμμιστούμε ακριβώς με τα όσα είπε η Επιτροπή Γεωργίας, πρόεδρος της. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε να εκφράσουμε και εμείς τις απόψεις μας. Και εμείς ήδη από την πλευρά της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουμε διοργανώσει μια ε, ε, συζήτηση με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά αυτή την ανακοίνωση, σε ό,τι αφορά την αποψήλωση των δασών ε, και νομίζω πως ε, αυτό καταδεικνύει ε, την μεγάλη μας ανησυχία από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά και τη σχέση ανάμεσα στην αποψήλωση αφενός και το εμπόριο αφετέρου. Νομίζω πως είναι πολύ θετικό εμείς, αυτέ οι επιτροπέ, δηλαδή, να συνεργαστούμε μαζί, η δική σας, Γεωργίας, και άλλες έτσι ώστε για παράδειγμα να φτάσουμε όχι υποχρεωτικά σε κάποιο ψήφισμα οτιδήποτε άλλο αλλά σε πολύ συγκεκριμένα μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα. Και αυτό το αναφέρω γιατί το άκουσα χθε από τον κύριο Τίμερμαντς από τη Νέα Υόρκη το ότι δηλαδή υπάρχουν δύο στοιχεία ή δύο τομεί για του οποίου ε, χρειάζονται νομοθετικέ προτάσει από την πλευρά τη Επιτροπή. Πρώτον, τα πλαστικά, για το οποίο δεν χωράει εμβολίο. Και από την άλλη πλευρά η αποψήλωση, η εισαγωγή δηλαδή προϊόντων που προέρχονται από αποψήλωση. Οπότε, ε, όταν ε, είδαμε εκείνη την διαφάνεια από την πλευρά της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, εκεί εγώ θα προσθέσε, προσέθετα συγγνώμη, ακριβώς νέες νομοθετικές προτάσεις από την Επιτροπή, από τον Επιτροπή. στο πλαίσιο του Green Deal. με βάση την νομοθεσία βέβαια για την ξυλία, για το φλέκτ και ούτω καθεξής θα δούμε τι ακριβώς θα προτείνουμε αλλά εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε για τέτοιου είδους νομοθεσία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι ώστε να προλιάνουμε το έδαφος προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το Green Deal. Ε, το τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να θέσω είναι το μέλλον των εμπορικών συμφωνιών. Δεν θα επανέλθω στο ζήτημα της Μερκοσούρ, αλλά ε, θα αναφερθώ σε μελλοντικέ, για παράδειγμα, όπως αυτή με το Βιετνάμ. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι υπάρχει εδώ ένα τεράστιο μέτωπο αποψήλωση στο Βιετνάμ. Το γνωρίζουν όλοι αυτό. Δηλαδή, αν ρίξει κανεί μια ματιά στι φωτογραφίε του δορυφόρου, βλέπει τη Μαλαισία, την Ινδονησία ε, και τώρα βλέπει και το Βιετνάμ και την Καμπότζη. Οπότε θα θέλαμε να ακούσουμε από την Επιτροπή ποιε είναι οι συγκεκριμένε προτάσει ή έστω οι δικλείδε ασφαλεία, αν θέλετε, τι οποίε έχει προβλέψει μέσα σε αυτή τη μελλοντική συμφωνία εμπορίου με το Βιετνάμ. Ακόμα κι αν τίθενται ε, ερωτήματα και μέσα στην ε, ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος από τις διάφορες πολιτικές ομάδες ως προς το ότι τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα, επιχειρησιακού αν θέλετε χαρακτήρα ε, και συγκεκριμένες ε, ε, δικλείδες ασφαλείας ή αυτά τα μέτρα δηλαδή που να διασφαλίζουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της Συμφωνίας των Παρισίων. Τι σημαίνει δηλαδή συγκεκριμένη εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων της Συμφωνίας των Παρισίων. Και τι για παράδειγμα σημαίνει όταν λέμε ότι δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά μια τέτοια δέσμευση από αυτή τη συμφωνία. Τι συμβαίνει σε εκείνη την περίπτωση. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, ένα πάνελ, μια ε, δημόσια θέση η οποία ε, υιοθετείται, αλλά από εκεί και μετά θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβαίνει. Και έτσι λοιπόν η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, δεν μιλώ εδώ δηλαδή, ε, δεν εκφράζω την προσωπική μου άποψη, αλλά μιλώ ως πρόεδρος της ομάδας περιβάλλοντος, τα περισσότερα λοιπόν μέλη επιθυμούν να υπάρξει μια κοινή δουλειά εδώ με την Επιτροπή, έτσι ώστε όχι να γίνει μια πολιτικού χαρακτήρα συζήτηση, αλλά προκειμένου να ξέρουμε πολύ συγκεκριμένε και ρεαλιστικέ απαντήσει στα ερωτήματα που μόλι έθεσα. Δηλαδή, ποιο αποφασίζει αν έχει εφαρμοστεί σωστά ή όχι μια τέτοια δέσμευση, τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν έχει εφαρμοστεί ε, μια τέτοια δέσμευση, αν θεωρηθεί πως δεν έχει εφαρμοστεί και ούτω καθεξής. Ε, και υπάρχει από δική μας πλευρά μια μεγάλη πλειοψηφία έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια νέα ισορροπία σε ό,τι αφορά το εμπόριο αφενός και την αποψήλωση ε, και το περιβάλλον γενικότερα αφετέρου. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας. Ε, δύο λεπτά ο καθένας. Η Χάιντι Χάουτελα έχει πρώτη το λόγο που ήταν η συγγήτριά μας ε, για το φλέκτη σε ό,τι αφορά το Βιετνάμ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως είμαστε τυχεροί που τον Ιούλιο τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε αυτό το σχέδιο δράσης και φυσικά του ασκήθηκε κριτική για το γεγονό ότι δεν ήταν ε, παρκώς ε, φιλόδοξο, αλλά νομίζω πως ε, βασίζεται στις κατάλληλε εκτιμήσεις. Και εδώ θα ήθελα να εστιάσω στο ζήτημα της ζήτησης. Ε, δηλαδή, πολλοί λένε ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράσει σε ό,τι αφορά την εισαγόμενη αυτή αποψήλωση, όπω λέγεται, αλλά αυτό ε, μπορεί να καταστήρει σαφές μόνο με την καλύτερη διαχείριση των αλυσίδων ε, παραγωγή αξία. Δηλαδή, εφόσον αυτέ είναι διαφανεί και γνωρίζουμε ακριβώ από πού προέρχονται τα εν λόγω προϊόντα στι εν λόγω χώρε εξαγωγή των προϊόντων δηλαδή κινδύνου που συνδέονται δηλαδή με κινδύνους αποψήλωσης. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει κατάλληλη νομοθεσία ε, για να ελέγχεται η δέουσα δεοντολογία. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ολοένα και περισσότερε επιχειρήσεις που εξάγουν αυτά τα προϊόντα ε, σε εμά ε, καλούν, θέλουν να υπάρχει νομοθεσία γιατί τελικά εκείνοι οι οποίοι αποφελούνται από τη μη ύπαρξη τέτοιων αυστηρών κανόνων είναι ακριβώς οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι διαφανείς. Οπότε ε, χαιρετίζω την πρόταση που έκανε και ο πρόεδρο ε, τη Επιτροπή Περιβάλλοντο να ξεκινήσουμε μια ευρεία συζήτηση στο Κοινοβούλιο για να δούμε τι είδου μέτρα νομοθετικού αλλά και μη χαρακτήρα προκειμένου να καταφέρουμε να σταματήσουμε το φαινόμενο αυτή τη αγόμενη αποψηλούση. Ε, και νομίζω πω θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτά τα προϊόντα υψηλού κινδύνου, αν θέλετε, σχέση με την αποψήλωση, όπως η ξυλία, για παράδειγμα, ε, και οικοκοφίνα και σε άλλα από εκεί και μετά, ενδεχομένω να χρειαζόμαστε ε, μια οριζόντιου χαρακτήρα νομοθεσία σε ό,τι αφορά την δέουσα διοντολογία σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση η νομοθεσία FLEG τα αναφέρθηκε εδώ επανελειμμένα και ε, νομίζω πω αυτό αποτελεί πραγματικά την κορονίδα, αν θέλετε, ε, τη ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθύνη από τι επιχειρήσει και σε ό,τι αφορά ε, το Βιετνάμ, ε, επιχαίρουμε το γεγονό αποτελεί αναπόσταστο τμήμα τη μελλοντική συμφωνία εμπορίου. Αλλά προτού υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία, θα πρέπει καταρχήν να ελέγξουμε πώ εφαρμόζει τι δεσμεύσει του το Βιετνάμ σε ό,τι αφορά ακριβώ την νομοθεσία FLECT. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε και εμεί από τη δική μα πλευρά τη Επιτροπή Εμπορίου. Ναι, και θα υπάρξει μια αποστολή μέσα στον Οκτώβριο από την πλευρά τη δική μα επιτροπή, στο πλαίσιο τη οποία θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στο FLECT. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξαιρετικό το κείμενο. Τρομάζει βέβαια όταν βλέπει κανείς ε, τις προοπτικές ε, εξαφάνισης του αρχαίου δάσους. Κάποιες ερωτήσεις. Το κείμενο μας λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 10% αποψήλωση σε παγκόσμιο επίπεδο για μια σειρά προϊόντων, καουτσού, καραβόστο κλπ. Συχνά στην Επιτροπή γίνεται μια στρέβλωση μεταξύ των λόγων και των έργων της Ένωσης. Μιλάμε για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Το Μαρκοσούρ, για παράδειγμα, έχει άμεσες επιπτώσεις στην αποψήλωση. Η καλλιέργεια της εθανόλης, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια τόνοι παράγονται στο Μερκοσούρ, αλλά ε, όταν λέμε ότι θα περάσει ελεύθερη Αθανόλη στην Ένωση, αυτό είναι ένα ευθύς, ευθύ μέτρο κινήτρου για την παραγωγή της. Η Ινδονησία από την άλλη. Ο ρυθμός εξαφάνισης του τροπικού δάσους στην Ινδονησία είναι ε, φρικτός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει επιπτώσεις η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Βιετνάμ. Μιλάμε για το φλεκτή. Η Κομισιόν μας λέει ότι αποτελεσματικό, ε, εύλογη ε, προθυμία, ωραία είναι αυτά, αλλά κάθε χρόνο έρχεται παράνομο, παράνομη ξυλία από το Λάος, την Καμπότζη, 300.000 κυβικά μέτρα ε, καμπο, ε, παράνομου, παράνομης ξυλίας από την Καμπότζη πέρασαν στην Ευρώπη μέσω Βιετνάμ. Αυτή είναι η πραγματικότητα των συμφωνιών ελεύθερης συναλλαγής. Κάτι άλλο που δεν συζητούμε πολύ. Το ευρωπαϊκό δάσος. Ωραία είναι αυτά που μας λένε. Μπράβο, αυξήσαμε την ε, δασική κάλυψη στην Ευρώπη. Να πούμε όμως ότι υπάρχει μία αλλαγή της δομής των δασών μας. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, αλλά αυτό σημαίνει και σε άλλες χώρες. Έχουμε σταδιακή υποκατάσταση ενός είδους ε, δέντρου, πεύκο, σε σχέση με παλιότερες ε, με παλιότερα δέντρα, βαλανιδιά, οξιά, ε, ε, οξιά λεύκα που σιγά σιγά εμφανίζονται νέα είδη που υποκαθιστούν τα παλιά στα δάση μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την περιγραφή της γενικής κατάστασης. Εγώ θα σταθώ στο θέμα της ετελικής σχέσης με, τα, με τις παραγωγούς χώρες. Η ιδέα του να έχουμε στη συνθήκη κάποιες συμβάσεις, ε, ε, κάποιες ρυθμίσεις, ε, μήπως κατά την, κατά άποψή μου είναι αρνητικό. Κατά την άποψή μου πρέπει να έχουμε αποτελεσματική εταιρική σχέση, partnership το λέμε, αλλά το να λέμε ότι η Ευρώπη πρέπει να δει τι κάνει η ίδια δεν είναι κακή γιατί και εμείς ε, ξεριζώνουμε δέντρα για να εκμεταλλευτούμε τη γη για γεωργικούς σκοπούς. Μήπως λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια εταιρική σχέση που συνοδεύεται από μια συμφωνία όπου λούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά την αναδάσωση και την βιώσιμη διαχείριση του δάσους. Γιατί το ένα ε, μπορεί να έχει εκμετάλλευση του δάσους χωρίς να καταστρέφεις το δάσος. Μπορεί να έχεις εκμετάλλευση δάσους με βιώσιμο τρόπο. Άκουσα σήμερα, διάβασα σήμερα στη Βύση ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε σήμερα στη Νέα Υόρκη πως μισό δις ε, δόθηκε σε κράτη για την καταπολέμηση της αποψήλωσης του δάσους. Από την Παγκοσμία Τράπεζα, από την Παγκόσμια από την Παναμερικανική Τράπεζα Επενδύσεων και από μία ΜΚΟ. Μήπως έπρεπε και η Ευρώπη να δημιουργήσει αυτή την πλήρη εταιρική σχέση για να κρατήσουμε τις επιφάνειές μας πράσινες για να αποφύγουμε την μετατροπή του δάσου σε γεωργική εκμετάλλευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σημαντική συζήτηση και ευχαριστώ και για την ανακοίνωση. Και είναι πολύ χρήσιμο το ότι έχουμε εκπροσώπους και από την Άγκρη και από την ΕΜΒΗ. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ξέρετε, είναι οι στόχοι, δεν αφορούν μία επιτροπή μόνο. Επίσης είναι σημαντικό όταν μιλάμε για αλλαγή του κλίματος και την απώλεια της, βιοπι... του κλίματος και την απώλεια της βιοποικιλότητας, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πώς οι μας, η δική μας παρέμβαση στο περιβάλλον έχει κάποιο αντίκτυπο στην αποψήλωση. Η ανακοίνωση δίνει τις δράσεις που χρειάζονται. Η Ένωση έχει κατανάλωση 10% σε παγκόσμιο επίπεδο προϊόντων που προέρχονται από την αποψήλωση. Ενδιαφέρον στην ε, έκθεση είναι η σημαντική αναφορά στην ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης και, στην, ε, και στο επίπεδο της ζήτησης και στο επίπεδο της προσφοράς. Είναι σημαντικό να προχωρήσει λοιπόν η Επιτροπή και θέλω να ρωτήσω υπάρχουν συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα πλάνα. Κοίταξα τα slides της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Βλέπω την κατάσταση ως έχει. Δεν βλέπω νέες δράσεις για την αντιμετώπιση της αποψήλωσης. Άκουσα ας πούμε για το Mercosur. Ε, μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι προϊόντα που εισάγονται από τη Βραζιλία δεν είναι προϊόν που προέρχεται από την αποψήλωση ή που σχετίζεται με την αποψήλωση. Μια τελευταία ερώτηση. Πολλές ΜΚΟ, Global Witness πρόσφατα, λένε ότι οι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί και οι τράπεζες χρηματοδοτούν έμεσα την αποψήλωση. Έχει κάποια νούμερα η Επιτροπή σχετικά. Έχει κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ.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 Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε την Επιτροπή. Νομίζω πω έρχεται στην κατάλληλη χρονική συγκυρία αυτή η συζήτηση, όπω και η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι πιο δυστάρεστο από το να βλέπει κανεί πυρκαγιέ ε, ανεξέλεγκτε. Ε, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή και τις ε, επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα και την χλωρίδα και την πανίτα και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να σταματήσουν τέτοιου είδους πυρκαγιές στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα παγκοσμίω. Και επίσης ε, όταν αναφερόμαστε σε εμπορικέ συμφωνίε με χώρε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα ακριβώ ότι υπάρχουν τέτοιε χώρε, για παράδειγμα στη Μερκοσούρ, η Βραζιλία ή το Βιετνάμ και η Ινδονησία, άλλου, όπου λαμβάνει η χώρα τόσο μεγάλη αποψηλωσία. Νομίζω πω θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι εάν συνεχίζεται η αποψήλωση σε αυτές τι χώρες δεν θα υπάρξει εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί και μετά, εφόσον συνεχίζεται αυτή η αποψήλωση, η εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από τις εν λόγω χώρες θα πρέπει να σταματήσει. Με αυτόν τον τρόπο θα ε, δώσουμε, θα περάσουμε το μήνυμα ότι θα πρέπει δηλαδή να αναλάβουν δράση αν θέλουν να υπάρξουν αποτελέσματα. Και βέβαια αυτά τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή πολλά μέλη είπαν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αποψήλωση, ειδικότερα ε, σε ό,τι αφορά ε, τα, ε, τα, τα δέτα τα οποία για παράδειγμα είναι σε εκείνες τις περιοχές όπου υπάρχουν δηλαδή παραδοσιακά. Ε, όπως και στη δική μου χώρα. Σε σχέση λοιπόν με τέτοιου είδους ε, χλωρίδα έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι ε, για, έως το 2030, αλλά θα πρέπει να ζητούμε συγκεκριμένα δεδομένα από τις εν λόγω χώρες ε, σε ό,τι αφορά το 2020, το 2021, το 2022, το 2023. Δεν έχει νόημα δηλαδή να παρακολουθούμε αυτές τις χώρες σε δεκαετή βάση. Σε σε βάση θα πρέπει να τις ε, παρακολουθούμε για να δούμε κατά πόσο επιτυχάνουμε συγκεκριμένη πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν να στήσω από τη νέα Επιτροπή να παρακολουθεί τα πάντα, να υποβάλλει εκθέσει και από εκεί και μετά να λαμβάνονται αποφάσει έτσι ώστε να ε, ασκούνται και κατάλληλε, να επιβάλλονται κατάλληλε κυρώσει σε περίπτωση μη πλήρωση αυτόν τον στόχο. Ναι, λέει ο πρόεδρο σε πολύ αυστηρέ ε, ε, προποθέσει. Κάτι Φαμπρέτ. Ευχαριστώ. Σημαντική συζήτηση αυτό το ζήτημα είναι ένα σημαντικό ζήτημα τόσο και για αυτήν εδώ την Επιτροπή αλλά και για άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές οπότε ελπίζω πως θα μπορέσουμε ε, ξεκινώντας αυτή την νέα θητεία να έχουμε μια ε, καλή συνεργασία μεταξύ μας. Αντίθετα με αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν, δηλαδή ο καθένας να προσπαθεί να προωθήσει αν θέλετε το δικό του χαρτοφυλάκιο ακόμα κι αν υπάρχουν ε, ιδεολογικές διαφορές ε, στις απόψεις μας, νομίζω πως τελικά όλοι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση σε σχέση με την αποξήλωση. Οπότε είμαι πραγματικά υπέρ της ε, συνεργασίας ανάμεσα σε αυτές εδώ τις επιτροπές που συμμετέχουμε σήμερα, αλλά και την ΕΚΟΤ και την ΑΦΕΤ και άλλες. Ένα δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω σχετίζεται και ερώτημα προς την Επιτροπή ως προς ε, τι ακριβώς κάνουμε σε, σε σχέση με τις αγωγές, για παράδειγμα όπως ε, στις χώρες της Μερκοσούλ. Είδαμε δηλαδή ε, τις απόψεις από την πλευρά του Ευρωσκηνού ότι δηλαδή εάν η Μερκοσούλ είχε μια συμφωνία μαζί μα αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα είχαν σημειωθεί πυρκαγιέ ε, στην Αμαζονία. Αυτό είναι μία άποψη, γιατί υπάρχει και άλλη άποψη, η οποία λέει ότι εάν δεν προβούμε στη σύναψη τη συμφωνία ε, με, τη, με το, τις της Μερκοσούρ, τότε θα καταφέρουμε να σταματήσουμε τις ε, πυρκαγιέ. Ε, παρουσιάζω λίγο απλουστευμένα και λίγο ακραία αυτέ τι απόψει, αλλά νομίζω πως καμία δεν είναι σωστή. Δηλαδή, το να πούμε ότι μέσα σε, στη σύναψη μια τέτοια συμφωνία θέτουμε και συγκεκριμένου στόχου σε ό,τι αφορά τις, ε, τη Συμφωνία των Παρισίων δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε την, ε, το πώ εφαρμόζεται ε, μια τέτοια συμφωνία και από εκεί και μετά θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προποθέσει πριν από την υπογραφή και την κύρωση μια τέτοια συμφωνία. Νομίζω πω αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το εξετάσει η Επιτροπή και σε αυτό θα πρέπει να πιέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και σε σχέση με τι σε σχέση με άλλε χώρε όπω από το Βιετνάμ, η Αυστραλία και άλλε. Και σε σχέση με αυτό το θέμα θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα. Κάτι δεν κατάλαβα. Αναφερθήκατε στη ρήτρα μη αναδρομή, το non-regression, δηλαδή ε, μια χώρα η οποία έχει συνάψει μια τέτοια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μαζί μας δεν επιτρέπεται να ε, μειώσει ε, τα δικά της πρότυπα, τα περιβαλλοντικά για παράδειγμα, εάν θέλει αύξηση του εμπορίου, δηλαδή για άλλους λόγους, για παράδειγμα αγροτικών προϊόντων εφοδιασμού με τρόφιμα θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει, να προβεί σε αναδρομή, δηλαδή να, μειώσει τα, τα, τα πρότυπά τη. Γιατί νομίζω πω κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Δηλαδή, στο πλαίσιο μια τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να είναι δυνατή να σε χαμηλότερα πρότυπα σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ. Μαντιλένα από την Επιτροπή, εσεί έχετε τώρα το λόγο για να δώσετε κάποιε απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι. Άστε Τσούμακερ, λοιπόν, από τη Γενική Διεύθυνση Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για τα σχόλια στου δύο πρόεδρου, Άγκρη και Έμβη κυρίω, και σε εσά. Είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κοινή προσέγγιση είναι χρήσιμη για να βρούμε την πιο σωστή προσέγγιση και μαζί όχι μόνο εμείς αλλά και η Γενική Διεύθυνση Trade και η DEVCO πρέπει να συνεργαστούν Από την οπτική μας λοιπόν και η Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει να εμπλέκεται στις συζητήσεις γιατί ό,τι κάνουμε πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι βοηθά και τις παραγωγούς χώρες. Το δάσος δεν το κόβουν γιατί έτσι θέλουν, γιατί χρειάζεται να επιβιώσουν. Πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε και εναλλακτικέ στις χώρες αυτές αν θέλουμε να έχουν μια σωστή αντιμετώπιση του δάσους. Ακούσαμε πολλά για το πώς μπορεί το εμπόδιο και το περιβάλλον να υποστηρίζει το ένα το άλλο. Κρίσιμο το ερώτημα που αφορά και τις υφιστάμενες συμφωνίες και τις, ε, την καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η κοινωνία των πολιτών σε κάθε χώρα για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τις δικές τους προοπτικές και να χρησιμοποιήσουμε το εμπόδιο όχι ως αυτοσκοπό, αλλά και για την προώθηση των υπόλοιπων στόχων της ε, ανάπτυξης. Αυτά τα πράγματα θέλουμε μαζί να τα δούμε. Πολλά ερωτήματα εύλογα για την αξιολόγηση των κανονιστικών και μη μέτρων. Συμφωνώ με όσους λένε ότι το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως επίγον και θέλουμε, ξεκινήσαμε την αξιολόγηση χωρίς καθυστέρηση. Απλώς να σας πω ότι αν θέλετε να κάνετε μία αξιολόγηση δικτύπου σωστά, όπως θέλουμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε νέα νομοθετικά κείμενα στα πλαίσια του European Green Deal μέσα σε 100 μέρες. Χρειάζεται καλή ανάλυση των πολιτικών που δούλεψαν καλύτερα, λαμβάνοντας υπόψη, το αναφέρατε αυτό, το γεγονός ότι η αλυσίδα της λειτουργίας του δάσους έχει κάθε μία διαφορετικές προτεραιότητες. Μιλήσαμε λοιπόν για το ρόλο του φλεκτ. Θέλουμε να δούμε και να σκεφτούμε πώς επηρεάζει αυτό. Ζητήματα πιστοτήπησης υποχρεωτικής επισήμανσης κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποφασίσει σαφώς τι χρειάζεται και τι όχι. Ένα συνδυασμό κατά πάσα πιθανότητα. Πάντως αυτό που θέλουμε είναι νομοθεσία που δεν θα μείνει στα χαρτιά, αλλά θα εφαρμόζεται αυτόματα και για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες ακόμα, χωρίς μεγάλους περιορισμούς, και για την παρακολούθηση της εφαρμογής. Στο πλαίσιο του EUTR θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται περισσότερη δουλειά για την εφαρμογή από τα κράτη και για τους πολίτες και τις αρχές. Αλλά οι αρχές είναι αυτές που πρέπει να δουν πολλές συμφωνίες και προσεγγίσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πολλοί αναφερθήκατε στο Βιετνάμ. Χάρηκα που άκουσα την πρόεδρο της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος να θέλει να, ότι θέλει να ταξιδέψει στο Βιετνάμ. Για μας είναι πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Έχει, έχουμε συμφωνήσει μια συμφωνία εταιρική σχέσης. Σε ό,τι αφορά το FLECT, ε, δείχνει ενδιαφέρον γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι, για μας τουλάχιστον είναι η εφαρμογή του φλεκτ στη χώρα παραγωγής, όχι στη χώρα αύξησης του, της ξυλίας. Και νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε. η συνάδελφος από το, τη trade θα σας Γενική Διεύθυνση Trade, θα σας μιλήσει και για την συμφωνία με το Βιετνάμ, αλλά ο στόχος είναι να εμποδίσουμε τις εισαγωγές παράνομης ξυλίας από το Βιετνάμ, ανεξάρτητα από το που είναι ο αρχικός τους, η αρχική τους προέλευση. Το θέμα είναι κυρίως εφαρμογή της νομοθεσίας στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ έχει νομοθεσία που απαγορεύει την, παρανομή, την χρήση και πώληση παρανομής ε, υλοτομημένης ξυλίας. Και αυτό δείχνει πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις εθελούσιες συμφωνίες. Η εμπλοκή των χρηματοδοτικών οργανισμών. Διαβάσαμε τη μελέτη αυτή, δεν έχουμε θέση προς το παρόν. Προς το παρόν. Η καθοδήγηση της χρηματοδότησης ωστόσο έχει πολλές δυνατότητες, ιδίως αυτό που θεωρούμε σημαντικό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση, διαφάνεια της χρήσης των κονδυλίων αυτό και αυτό είναι κάτι που εμείς θα κυνηγήσουμε. Παρατηρητήριο. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία θέση σε λειτουργία. Συνεχίζεται η προπαρασκευαστική δουλειά. Η παρακολούθηση της αναδάσωσης, από όσο ξέρω, προφανώς είναι μέσα στις αρμοδιότητες του παρατηρητηρίου και πληροφορίες και από ΜΚΟ στις χώρες παραγωγής. Το σημαντικό είναι να διαφέρουμε τις πληροφορίες αυτές σε όλους και στις χώρες παραγωγής. Δεν θυμάμαι αν υπήρχαν δώσω Δίνω το λόγο στη συνάδελφο. Ε, και άλλες απαντήσεις. Ε, και άλλες απαντήσεις είναι ένα θέμα με πολλές πτυχές. Πρέπει να το δούμε πολλές φορές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, καταρχάς το θέμα της δεύτερης επιμέλειας. Έχει πολλέ πτυχέ. Έχουμε τακτικές συνεδριάσει με υπηρεσίες κομισιών, τη Γενική Διεύθυνση Grow, η οποία συντονίζει. Η Γενική Διεύθυνση Justice ε, κάνει μια μελέτη αντικτύπου, πολύ σημαντική για, σημαντική για την αλυσίδα ανεφοδιασμού, για να δει τι ανάγκες έχουμε για το due diligence. Η FISMA ασχολείται με την νομοθεσία που δεν είναι οικονομική φύσεως. Η DEFCO είναι δραστήρια επίσης η Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, επίσης το διεθνές επίπεδο, όπου έχουμε δράσεις ε, σε πολλά επίπεδα. Πολλοί εμπλέκονται. Σωστά λέτε ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να τα καταφέρουμε. Να ξεκινήσουμε το Βιετνάμ τώρα. Χαιρόμαστε που θα πάτε στο Βιετνάμ. Το Μάιο είχα πάει για δράσεις ε, εφαρμογής για το τσάι. Συζητήσαμε και το ΦΛΕΚ τότε. Ε, έχουμε ξεκινήσει έτσι μια σχέση με τους Βιετναμέζους. Ε, συζητήσαμε και εργασιακά θέματα. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η χώρα. Κοιτάζει σοβαρά τις διεθνείς δεσμεύσεις για θέματα περιβάλλοντος επίσης, κλίματος, φλεκτ και για τα εργασιακά θέλουν να δουν τι δράσεις μπορούν να λάβουν για να εφαρμόσουν τις μελλοντικέ συμφωνίες και αυτά που, αυτές που ήδη υπάρχουν στα πλαίσια του φλερτ. Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι το ποιος αποφασίζει. Τι είναι ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή μιας συμφωνίας. Να μην σας δώσω μια νομικήστικη απάντηση. Ε, ασχολούμαστε στα πλαίσια του πάνελ με τη, για τη συμφωνία με την Κορέα. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή το πάνελ αυτό. Πριν φτάσουμε στο πάνελ όμω οτιδήποτε κάνουμε ε, έχει ένα στάδιο παρακολούθηση ε, της εφαρμογής με τον εταίρο της Συμφωνίας Μπορείου. Και κάθε φορά του λέμε εφαρμόζεται το ΧΙΠΣΙΖ. Το συζητάμε δηλαδή. Αλλά τελικά όμω, υπάρχει και ένα πάνελ το οποίο αποφασίζει τελικά αν υπάρχει εφαρμογή σωστή ή όχι. Ε, Επίσης, κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις με τους εταίρους μας, τι σημαίνει το Παρίσι, η Συμφωνία του Παρισιού, ε, οι συμφωνίες ε, ILO, ε, τις ε, διμερείς συμφωνίες τις ομαδόμες πολυμερείς συμφωνίες. Ο ILO ε, θα σας πει ότι υπάρχουν διάφορες επιτροπές που εφαρμόζουν τις διάφορες ε, διατάξεις. Εμείς συνεργαζόμαστε ω Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, γιατί έχουμε και τη δική μας ερμηνεία για ότι είναι αποτελεσματική εφαρμογή. Έχουμε και διάφορες δομές ε, παρακολούθησης, ε, εταιρική σχέση, σημαντική. Το 10% της κατανάλωσης είναι από εμά. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το 90% καταναλώνουν άλλοι από μόνοι μας δεν θα πετύχουμε τίποτα. Αν δείτε την αλυσίδα ανεφοδιασμού, ας δούμε το κακάο, ας πούμε, που είναι κοντή αλυσίδα. Οι περισσότερες όμως αλυσίδες είναι περίπλοκες και περνάνε τα σύνορα. Ε, έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, άρα πρέπει να συνεργαστούμε με πολλές χώρες. Να χτίσουμε συμμαχίες για να τα καταφέρουμε. το αποτύπωμά μας, το μεριδιό μας στην κατανάλωση. Τα τελευταία πέντε χρόνια, με τις εφαρμογές TST, εστιάσαμε στη, στα εργασιακά και τα τελευταία δύο-τρία χρόνια στο κλίμα. Δεν θυμάμαι τα τέσσερα χρόνια που είμαι εδώ, να, πέρα από το να θέτουμε θέματα, δεν σκεφτήκαμε Πώ θα εφαρμόσουμε αυτέ τις διατάξεις, α πούμε, το Mercosur και διάφορες διατάξεις που δεν εφαρμόζονται, δεν έχουμε σκεφτεί πώ θα τις ε, καταστήσουμε πιο αποτελεσματικέ. Έχουμε μια ευκαιρία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο ε, εφαρμογή με σχέδια δράση, ε, συζητήσει σε πολυμερή φόρουμ, να εξηγήσουμε τις δικές μας νομοθετικές εξελίξεις στους εταίρους. Υπάρχουν νομοθεσία που μπορεί να τους αρέσει περισσότερο ή να νομοθεσία που να μην του αρέσει. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο έχει διάλογο. Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία με το Μερκοσούρ. Αν κοιτάξετε συνολικά τις διατάξεις που συνδέονται με τα βάση, μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα. Επίσης, οι στατιστικές. Δεν ξέρω ποιο έχει έρθει από πλευρά Κομισιόν, αλλά δούμε το Βόϊο. Ε, εισαγωγέ βόιου Είναι 200.000 τόνοι. Με βάση ε, δασμού ε, ύψου 40 με 45%. Έχουμε μια ποσόστοση 99.000 τόνους. Το μισό από αυτό έχει δασμούς 7,5%. Δεν περιμένουμε δηλαδή οι εισαγωγέ να αυξηθούν. Περιμένουμε μάλλον ότι αυτές οι εισαγωγές θα ενσωματωθούν στην ποσόστοση και θα τις απορροφήσει η ποσόστοση. Επίσης, σε σχέση με την αποψήλωση, η ποσόστοση που έχουμε το Μερκοσούρ είναι το λιγότερο το 1% της α, παραγωγής Βραζιλίας. Η ποσόστοση που έχουμε εμείς, δηλαδή η επίπτωση που θα έχει στην αποψήλωση το, της ποσόστοσή μας του βόλου είναι μικρή, έτσι. Δεν πρέπει να, να μην τονίσουμε βέβαια και τη σημασία, αλλά πρέπει να δούμε ας πούμε, τη σχετική σημασία που έχει το βόλιο σε αυτή τη συζήτηση, η παραγωγή Εν συνεχεία. Λύσεις μέσω της εμπορικής πολιτικής φυσικά θέλουμε να συνεισφέρουμε. μερικές φορές ε, αποδίδονται πράγματα στην εμπορική πολιτική που δεν είναι σωστά κατά ανάγκη. Φυσικά συνεισφέρουμε και φυσικά συνεργαζόμαστε και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στον τομέα τη δεούσα επιμέλειας. Αν υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία που προκύπτει από εκεί, δεν έχει να κάνει με την εμπορική πολιτική. Φυσικά είναι σημαντική, συνεισφέρουμε όσο μπορούμε, αλλά αν εσά είναι ας πούμε θέμα τη εμπορική πολιτική, εντάξει το δέχομαι. Ε, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε το αν θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική διάταξη για τη δέωση επιμέλεια. Ε, νομίζω ότι η επόμενη Κομισιόν θα αντιμετωπίζει, αντιμετωπίσει αυτή τη συζήτηση πολύ έντονα. Πράσινη Συμφωνία. Δεν έχουμε ένα πλήρες πλαίσιο αυτής της Πράσινης Συμφωνίας. Στην προετοιμασία είμαστε. Η νέα Κομισιόν σε 100, μέρες, σε 100 μέρες θα παρουσιάσει κάτι για αυτή την πράσινη συμφωνία, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Επί... Έπειτα πολύ σωστό είναι ότι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε πράξη αυτά που λέμε. Ε, φυσικά πρέπει να τα κάνουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Για τη ρήτρα μη επαναχώρησης, που είναι αμεληταία δεν ξέρω αν κατάλαβα την ερώτηση. Δεν ε, υπερβάλλει, δεν ε, έχει πρωτοκαθεδρία σε σχέση με την νομοθεσία. Ε, μιλάμε για εμπορικές συμφωνίες. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορείτε να μειώσετε τα, ε, τα πρότυπά σας για να προσελκύσετε τους, α, τις επενδύσεις και το εμπόριο. Δεν θα πρέπει η εμπορική συμφωνία να οδηγεί σε υποβάθμιση των προτύπων. Δεν θα Πρέπει να προωθείτε το εμπόριο με τρόπο που να υποσκάπτει τα πρότυπα. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για τη μελέτη αντικτύπου και το αν μειώνουμε τα πρότυπα της μελέτης αντικτύπου ώστε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις στην εξωτερική βιομηχανία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει η εμπορική συμφωνία. αλλά τίποτα πέραν αυτού. Αλλά ας δούμε και λίγο την απόδειξη των όσων λέμε. Ε, όχι λόγια μόνο, και αποδείξεις. Σούπερ, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Όπως είπε και η Ματλέν, δεν το συζητάμε το θέμα αυτό για τελευταία φορά. Φυσικά, ο πρόεδρος της Επιτροπής ΔΕΒΕ είχε προσκληθεί σήμερα αλλά δεν παρέστη, δεν μπόρεσε να έρθει. Και στην ε, τελευταία κοινοβουλευτική θητεία, ε, εμείς, δεν θέλουμε να, εμείς προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε την ιδέα του ότι η κάθε επιτροπούλα εργάζεται στο δικό της πεδίο. Θέλουμε συνεργασία με πολλές επιτροπές. Κλείσαμε εδώ το σημείο 9 και θα πάμε στο 10. Νέες εξελίξεις στην έρευνα για το εμπόριο σε υπηρεσίες και κρατικές προμήθειες. Το εμπόριο φυσικά σημαντικό σημείο, αλλά και η σύναψη δημοσίων προμηθειών είναι πολύ σημαντικό. 13 με 15% του ΑΕΠ ε, είναι οι προμήθειες αυτές. Προμήθειες και υπηρεσίες είναι σημαντικές για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μας. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον βασικό οικονομολόγο για το ε, εμπόριο, Λουσιάν Σερενάτ, που είναι Σελνάτ. Εδώ είναι. Θα μας κάνει μια παρουσίαση για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, δηλαδή για το ενδιαφέρον που δείχνετε για δύο πολύ σημαντικά αλλά και περίπλοκα ζητήματα της χάραξης εμπορικής ε, πολιτικής, ε, δηλαδή ε, το ζήτημα των υπηρεσιών αλλά και των προμηθειών. Όπως είπε και ο κύριος Λάγκε, είναι εξαιρετικά σημαντικά από οικονομική άποψη ε, ζητήματα και είναι εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα και σε ό,τι αφορά και την διαπραγματευτική μας ατζέντα. Σήμερα εγώ θα ήθελα να κοινοποιήσω και να μοιραστώ μαζί σας ε, τα αποτελέσματα ή και τα επερχόμενα αποτελέσματα ε, κάποιων πρωτοβουλειών που ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρχίζουν τώρα να αποφέρουν καρπούς. Ε, και μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και τη διαπραγματευτική ατζέντα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτά τα θέματα, γιατί είτε είστε νέο είτε παλαιό μέλος, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεστε την εξαιρετική σημασία αυτών των δύο ζητημάτων. Και τα νέα αναλυτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα ε, έχουν ακριβώ το στόχο να καταστήσουν ευκολότερη τη ζωή και τη δική μα, τη Επιτροπή, αλλά και τη δική σα, έτσι ώστε να αντιλαμβανόμαστε όλοι καλύτερα τι ακριβώ συμβαίνει. Να περάσουμε στην πρώτη διαφάνεια ω προ το τι ακριβώ θα σα παρουσιάσω, τι δηλαδή καλούμαστε να αντιληφθούμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τι διαπραγματεύσει, σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τι υπηρεσίε, αυτό πρέπει να αντιληφθείτε ότι παρά ε, της ε, διαπραγματεύσεις 25 ετών σε ό,τι αφορά το τομέα των υπηρεσιών δεν είχαμε ακόμα δεδομένα μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τις κύριες παραμέτρους ε, ε, σε ό,τι αφορά ακριβώς τον τομέα των υπηρεσιών και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα είδη υπηρεσιών, τα τα, τα είδη παροχής των υπηρεσιών. Άρα λοιπόν αυτό που θα σας πω εδώ σήμερα είναι ότι ακριβώς μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων τώρα για πρώτη φορά έχουμε τα απαλέτα αναλυτικά εργαλεία έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι τα δεδομένα σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες και προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις έχοντας τις προτεραιότητές μας και γνωρίζοντας τι συμβαίνει ακριβώς ειδικότερα. Εδώ αντιλαμβανόμαστε ε, την, ε, το, το είδος της παροχής υπαριθμών 3, το οποίο βασίζεται στι άμεσες ξένε επενδύσει και είναι εξαιρετικά σημαντικό ο τομέα. Και από εκεί και μετά έχουμε ε, το, τον τρόπο παροχή υπαριθμών 1, το MOD 1, που αναφέρεται στι ψηφιακέ υπηρεσίε και αντιλαμβάνεστε γιατί αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο η σημασία αυτών των ψηφιακών υπηρεσιών. Τώρα λοιπόν έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα για αυτούς ε, τους ε, τρόπους παροχής. Ε, και από εκεί και μετά κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι η σχέση ανάμεσα στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Δηλαδή, ακριβώς επειδή ο τομέα τη μεταποίηση είναι πολύ σημαντικό σε μια σειρά από κράτη-μέλη, θα πρέπει να υπάρχει και ένα αντίστοιχο επίπεδο υπηρεσιών που θα προωθεί στι αγορέ τα εν λόγω προϊόντα. Και σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες η κατάσταση σχέση με τα δεδομένα είναι χειρότερη γιατί παρότι υπήρχαν κάποια δεδομένα έστω σε ό,τι αφορά και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση στις ε, κρατικές ε, συμβάσεις δεν είχατε δει ποτέ τίποτα μέχρι τώρα και αυτό γιατί ακόμα δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα στη διάθεσή μας σε ό,τι αφορά τις ε, διεθνείς ε, κρατικές ε, συμβάσεις ε, και τώρα στις 13 Νοεμβρίου σας καλώ να συμμετάσχετε στην πρώτη δημοσίευση την οποία θα κάνουμε σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτά τα δεδομένα δηλαδή τις συμμετοχές των επιχειρήσεων σε διαδικασίες κρατικών συμβάσεων, κρατικών διαγωνισμών παγκοσμίω και από εκεί που δεν είχαμε καθόλου ε, δεδομένα τώρα έχουμε 38 εκατομμύρια επιμέρους δεδομένα σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, ε, κρατικές συμβάσεις. Να ξεκινήσω λοιπόν με την εξέταση του καταρχήν του τμήματος των υπηρεσιών και του, των τρόπων παροχής που αποτελεί ένα είδος έτσι, τεχνική ορολογία, αν θέλετε, σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να σα εξηγήσω το γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα στοιχεία η τρόπη παροχή. σω λοιπόν να έχετε δει ε, στι ειδήσει ε, το ζήτημα ε, γύρω από τον Τόμα Κουκ και το γεγονός που αντιμετωπίζουν ε, ε, χιλιάδες πολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτες χώρες ε, και αυτό ακριβώς βασίζεται στις ε, διεθνείς ε, υπηρεσίες. Δηλαδή κάποιος πάει στην αλλοδαπή ούτως ώστε να απολαύσει υπηρεσίες, υπηρεσίες εκεί για να βγάλει μια φωτογραφία για παράδειγμα τον πύργο των Άιφελ ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό σημαίνει ένα συγκεκριμένο είδος παροχής υπηρεσίας. Τώρα αν πάει κάποιος στην Καλιφόρνια για να κατασκευάσει βίλες για πολύ επιτυχημένους εργαζόμενους στο Silicon Valley Ω Δανό αρχιτέκτονας, αυτό το είδο παροχή τη υπηρεσία θα ήταν ένα ένας τρόπος παροχής που αντέχει στον τρόπο υπαριθμών 3. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικά είδη παροχή υπηρεσία, διαφορετικά είδη υπηρεσιών, τα οποία υπόκειται και σε τελείω διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια. Απλώ δεν είχαμε κανένα είδους πληροφορίε μέχρι τώρα ω προ τη σημασία των επιμέρους τρόπων και τι ακριβώ συμβαίνει στο ε, παγκόσμιο εμπορικό επίπεδο. Άρα λοιπόν αυτό που κάναμε ήταν, και θα δείτε και συγκεκριμένα αποτελέσματα στην επόμενη διαφάνεια, ε, να συνεργαστούμε με την Eurostat και με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εκπονήσουμε τα σχετικά δεδομένα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Δημιουργήσαμε λοιπόν μία ανάλυση των υπηρεσιών για κάθε κράτος μέλος, για κάθε τομέα υπηρεσίας ε, σε ό,τι αφορά τους κύριους προορισμούς. Όμως ε, ε, το απαιτούμενο ήταν από την πλευρά της Eurostat να συμμετέχουν τα ίδια τα κράτη-μέλη, αλλά μόνο το ίμιση των κρατών μελών ήταν διατεθειμένα να βοηθήσουν την Eurostat, γιατί ε, στο σε αλλά και αλλού σε πολλά άλλα φόρα. αναφέρθηκε ότι ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί ένα τομέα πολιτικής υψηλής προτεραιότητας. Αλλά όταν θέλουμε να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μπορέσουμε να θέτουμε και τι κατάλληλε προτεραιότητε, δεν έχουμε τα απαραίτητα δεδομένα στη διάθεσή μα για να το κάνουμε. Οπότε θα ήθελα να περάσετε αυτό το μήνυμα και στι δικέ σα χώρε, στου συναδέλφου σα και να του ρωτήσετε. Συμμετείχατε σε αυτή την προσπάθεια, βοηθήσατε την Eurostat να συγκεντρώσει τα σχετικά δεδομένα έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε και τι αποφάσει μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ένα ακόμα ε, στοιχείο το οποίο ε, δεν το έχουμε στη διάθεσή μα ή το έχουμε μόνο ελληπώ, είναι αυτό που αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δηλαδή συχνά αυτό ο τομέα των υπηρεσιών παρουσιάζεται ω ένα τομέα ε, του οποίου τα ωφέλη απολαμβάνουν μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αυτό ισχύει σε κάποιου τομείς αλλά σε άλλου όχι. Και πάλι θέλουμε να έχουμε περισσότερα δεδομένα για να δούμε τι ακριβώ μπορούμε να κάνουμε παραπάνω προκειμένου οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να μπορούν να ε, εποφεληθούν από την παγκόσμια αγορά υπηρεσιών και πάλι εδώ είχαμε ελάχιστα δεδομένα και λίγα τα κράτη-μέλη τα οποία μας βοήθησαν με την παροχή δεδομένων. Πάντως, πρωτού επιστρέψω στο ζήτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να σας πω ότι το ότι όταν θα βλέπουμε να υπάρχει μια προτινόμενη συμφωνία ε, υπηρεσιών, αυτό που λέγαμε παραδοσιακά ήταν ότι ε, οι εξαγωγές προϊόντων ε, και γενικότερα το εμπόριο προϊόντων από ό,τι υπηρεσίες, αλλά εάν προσθέσουμε όλα τα είδη ε, παροχής των υπηρεσιών, τα διαφορετικά είδη υπηρεσιών, δηλαδή τον τρόπο 1, τον τρόπο 3 και όλους τους άλλους, ουσιαστικά διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει πολύ περισσότερες υπηρεσίες από ό,τι προϊόντα. Η αξία δηλαδή των εξαγόμενων υπηρεσιών της Ένωσης υπερβαίνει την αξία ε, των ε, εξαγόμενων προϊόντων. Εδώ αν δείτε άλλο είδος στατιστικές θα δείτε ότι παρουσιάζουν λαθασμένη εικόνα, εσφαλμένη εικόνα. Αλλά θα σας δείξω και πιο συγκεκριμένα στοιχεία ε, σε λίγο, σε ό,τι αφορά και τα επιμέρους κράτη-μέλη και σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ σας δείχνω κάποια κράτη-μέλη με μικρομεσαίε επιχειρήσεις και βλέπετε ε, πόσο διαφορετική είναι η κατανομή, η διάρθρωση αν θέλετε του τομέα των υπηρεσιών σε διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή στην Ιρλανδία βλέπουμε ότι κυριαρχούν οι μεγάλε επιχειρήσει εκεί στον ε, παροχή των υπηρεσιών. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ονομαστικά αυτέ τι επιχειρήσει οι οποίε ε, κυριαρχούν εκεί. Αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες ε, χώρε Ανατολική Ευρώπη, για παράδειγμα η Εστονία, η Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο, όπου οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι εκείνε που καταλαβαίνουν το μεγαλύτερο μέρο των εξαγόμενων υπηρεσιών προ την Ε, συχνά δηλαδή πρόκειται για startups ή για επιχειρήσεις οι οποίες ε, άρχισαν να δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά καθώς συστάθηκαν από νέους τελειόφυτους. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να παρέχουμε υποστήριξη και σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα στην επόμενη διαφάνεια θα ήθελα να σας εξηγήσω ε, πώς έχουμε εξαγάγει τις βέλτιστες πρακτικές μας σε ό,τι αφορά αυτή τη συγκέντρωση των δεδομένων ε, ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Καταρχήν βασιστήκαμε, όπω σα είπα, στη διαδικασία τη Eurostat, αλλά αυτό δεν θα ήταν ε, επαρκέ αν δεν είχαμε δηλαδή και τι ε, κατάλληλε πληροφορίε από του εμπορικού μα εταίρου. Γι' αυτό λοιπόν πείσαμε την γραμματεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, έτσι ώστε να υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων με τα ίδια χαρακτηριστικά, με τα ίδια δηλαδή δεδομένα για 200 χώρε και καλύπτουμε τους ίδιους ε, ε, κλάδους όπως αυτοί καλύπτουν στη Συμφωνία GATS ε, για, για τις υπηρεσίες και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε δυναμικά σε βάθος χρόνου την εξέλιξη των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, αν εξετάσουμε για παράδειγμα τρεις χώρες που μας ενδιαφέρουν μέσα στα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την, τις υπηρεσίες, για παράδειγμα ε, την Ινδία ή την Ιαπωνία ή τις ΗΠΑ, χωρί αυτά τα δεδομένα δεν θα μπορούσαμε να δούμε ποια είναι η σχετική σημασία της ε, κάθε μίας από αυτές τις τρίτες ε, χώρες. Για παράδειγμα, αν δούμε για παράδειγμα ποιο είναι ο συνολικός, η συνολική αξία των υπηρεσιών που εξάγει η Ινδία και το συγκρίνουμε με τον όγκο της αξίας υπηρεσιών που εξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε ότι δεν είναι τόσο σημαντική η Ινδία και επίσης ε, τα δύο τρίτα των εξαγωγών ε, υπηρεσιών της Ινδίας γίνονται με, ε, της ψηφιακής οδού, ενώ αντιθέτως αυτή η εξαγωγή υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μόνο κατά το 1 τρίτο μέσω της ψηφιακής οδού. Οπότε αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να καταλάβουμε αν κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και αν είμαστε έτοιμοι για την τεχνολογική επανάσταση η οποία ακριβώς συντελείται με τις ψηφιακές εξέλιξεις. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ δυνατότητες λεπτομερούς χαράκτη τη ε, πολιτική λαμβάνοντα υπόψη αυτά τα επιμέρου ενδεδομένα. Άρα λοιπόν αυτά είναι κάποια παραδείγματα για τα στοιχεία τα οποία πλέον έχουν στη διάθεσή του οι αρμόδιοι για παράδειγμα για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτική, ε, σε ό,τι αφορά μάλιστα και επιμέρου τομεί, επιμέρου είδη υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε, υπηρεσίε τηλεπικοινωνιών ε, και ούτω καθεξή. Δηλαδή 58 επιμέρου κλάδους υπηρεσιών σε 200 χώρε σε αυτή τη βάση δεδομένων του ε, ΠΟΕ. Αυτό λοιπόν ήθελα να σα εξηγήσω ότι από ουσιαστικά μηδενικά δεδομένα που είχαμε σε ό,τι αφορά την χάραξη της πολιτικής μας γιατί ουσιαστικά ε, τα είχαμε αθρηστικά, αλλά όχι ξεχωριστά σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε. Τώρα έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα στη διάθεσή μα. Τώρα θα ήθελα να περάσω στο δεύτερο τμήμα, ή μάλλον προτού το κάνω, ε, θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην σημασία που έχει η σχέση ανάμεσα στη μεταποίηση αφενό και τι υπηρεσία αφετέρου. Είπαμε ότι προβαίνουμε στην πώληση υπηρεσιών, για παράδειγμα, για ψηφιακών διάβλων ή άλλων, αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχουμε μια ιδιαίτερα, ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο μεταποίηση, πρέπει να συνοδεύεται από τι ε, κατάλληλε υπηρεσίε ε, services in box όπως λέγονται, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική τεχνολογία που περιλαμβάνεται σε ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο τέτοιο αυτοκίνητο, ε, μια τεχνολογική συσκευή δεν θα είχε ε, την ίδια αξία αν δεν συναδευόταν από το κατάλληλο λογισμικό. Άρα λοιπόν, εδώ οι λειτουργίε αυτέ που προστίθενται μέσα από αυτέ τι υπηρεσίε είναι που δίνουν την αξία σε αυτό το προϊόν. Είτε πρόκειται για το μηχανολογία, είτε πρόκειται για το σχεδιασμό, για οικολογικό σχεδιασμό. Για παράδειγμα, ένα προϊόν το οποίο καταναλώνει ε, λιγότερη ενέργεια ή έχει λιγότερε εκπομπέ. Όλα αυτά δηλαδή η αξία του οικολογικού σχεδιασμού πρόκειται για παράδειγμα παροχή οι Αν θέλουμε, για παράδειγμα, να έχουμε πολιτικέ οι οποίε προστατεύουν τον περιβάλλον, τότε πάντοτε έχουμε να κάνουμε υπηρεσίε τέτοιου είδου οι οποίε περιλαμβάνονται, σωματώνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ε, προϊόν. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα τρόπο με τον οποίο με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να διασφαλίζουμε το πώ αυτέ οι τεχνολογικέ εξελίξει συνάδουν και με του εμπορικού κανόνε. Γιατί είναι περίπλοκοι αυτοί οι κανόνε. Έχουμε ε, την ΚΑΤ σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, την ΚΑΤ σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε ε, ε, και δεν υπάρχει μια σχέση ανάμεσα σε αυτέ τι συμφωνίε όπω συμβαίνει για παράδειγμα εδώ ανάμεσα στα διαφορετικά κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε. Ενώ αντιθέτω αυτή η σχέση και οι συνέργειε υπάρχουν κάθε φορά που κατασκευάζεται ένα τέτοιο προϊόν που περιλαμβάνει αυτέ αυτές τις υπηρεσίες. Άρα λοιπόν αυτό ήταν ένα ακόμα σημαντικό μήνυμα από το οποίο ήθελα να σας περάσω και βλέπετε εδώ 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας οι οποίες εξαρτώνται ακριβώ από αυτές τις συνέργειες που δημιουργούμε ανάμεσα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. briefly uh, to you. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο θέμα που θέλω τονίσω. Όπως σας είπα, οι κρατικές προμήθειες είναι μεγάλο κομμάτι κάθε οικονομία τη αναπτυσσόμενες 15 με 20% του ΑΕΠ κάθε χώρα. Τακτικά προσπαθούμε να εισάγουμε κανόνες που θα διέπουν την, τις κρατικέ κρατικές με, μέσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ που προσπαθεί να δημιουργήσει ισότιμο πεδίο λειτουργίας τόσο ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να μπορούν να κερδίσουν μια προμήθεια αν έχουν την καλύτερη προσφορά. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, πες ότι οδηγεί σε, σε έναν αυτοκινητόδρομο με μεγάλη ταχύτητα χωρίς φώτα. Ε, κάνουμε, οι διαπραγματευτές μας κάνουν πολύ καλή δουλειά χωρίς να έχουν φως να τους καθοδηγεί. Ε, δεν είχαμε στοιχεία να παρακολουθήσουμε, ενώ είχαμε κανόνες. Ξεκινήσαμε λοιπόν μία αναλυτική πρωτοβουλία που λέγεται IPPI, International Public Procurement Initiative, μην το παιδεύουμε το IPI που συζητείται στο το μέσο διεθνών προμηθειών, είναι αναλυτικό μέσο αυτό που σας λέω εγώ. Μαζεύουμε στοιχεία από τις μεγάλες χώρες, βλέπετε Κίνα, Ινδία, Βραζίλ, Ινδονησία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ταϊλάνδη, ΙΠΑ και Καναδά, με δημόσια στοιχεία διαθέσιμα δηλαδή στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη Βραζιλία ή στην Αυστραλία και προσπαθούμε να δούμε συχνά με τους κανόνες διαφάνειας ποιοι κέρδισαν μια προμήθεια, πού βρίσκεται η εταιρεία, πώς την κέρδισαν. Με αυτή τη μεθοδολογία έχουμε κάνει μια βάση δεδομένων με 13 εκατομμύρια συμβάσεις από τις χώρες αυτές και από τις 38, συγγνώμη, αυτές 38 ε, εκατομμύρια ε, συμβάσεις βλέπουμε πόσες τις κέρδισαν ντόπιε εταιρείε, πόσες ευρωπαϊκές, πόσες ιαπωνέζικες κλπ. Ούτω ώστε να έχουμε μια σωστή συζήτηση, πιο οθολογική συζήτηση για τη σημασία των κρατικών προμηθειών και της διεθνούς διάστασης τους. Εδώ σας δίνω μια εικόνα του έργου ξεκινήσαμε από το 0 μέχρι τα 38 εκατομμύρια με μια νέα μεθοδολογία συλλογής δεδομένων που έχει μόνο δημόσια διαθέσιμα στοιχεία. Δημιουργούμε ένα παγκόσμιο στάντα του, της έννοιας δημόσιου αγαθού και μετά μας ακολούθησαν και ο ΩΣΑ για παράδειγμα και, άλλες, και άλλοι διεθνείς οργανισμοί προσπαθώντας να δουν με έναν πιο εναρμονισμένο ορισμό. Η τελευταία διαφάνεια Έχουμε, όπως σας είπα, μια μεγάλη συνάντηση 13 Νοεμβρίου. Νομίζω έχετε προσκληθεί. Ελπίζω ότι θα έχουμε αρκετό χώρο να σας υποδεχθούμε όλους με συγκεκριμένα πολιτική στοιχεία της πρωτοβουλίας με βάση, στοιχεία, με βάση δεδομένα, μια εικόνα της πρωτοβουλίας με βάση δεδομένα και διαθέσιμα δεδομένα. Αυτό, αυτό είναι καινούριο. Για παράδειγμα, όταν κάναμε τι ε, διαπραγματεύσεις του Καναδά δεν είχαμε στοιχεία. Τώρα με την Αυστραλία έχουμε. Τα στοιχεία του Καναδά βέβαια τα χρησιμοποιούμε τώρα για να κάνουμε παρακολούθηση της ε, διαδικασία σήμερα. Επίση, ενισχύουμε και τη διαφάνεια, κάτι που είναι θετικό γιατί μιλάμε για τελικά για κρατικό ιδιωτικά κονδύλια, για, για λεφτά των πολιτών. Άρα η παρακολούθηση του που διατίθενται αυτά τα χρήματα είναι πάντα χρήσιμα και χρήσιμη και ε, θετική. Εντυπωσιακά λέει ο πρόεδρος, 38 εκατομμύρια συμβόλαια. Θα έρθουμε βέβαια στις 13 Νοεμβρίου. Κύριε Μπουζούα, ε, μάλλον έχετε ερωτήσεις. Τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω. Πρώτον, ευχαριστώ για την εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα εισήγηση. Η Κομισιόν χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα για την εκμετάλλευση των υπηρεσιών τη. Εγώ, όπως σας είπα, ήμουν υπουργό υπεύθυνο για τις εξαγωγές στη Φλάνδρα. Συχνά δεν είχαμε στοιχεία για τις εξαγωγές. Είχαμε στοιχεία για τις εξαγωγές αγαθών, αλλά όχι για τις υπηρεσίες. Δεν είχαμε αρκετά στοιχεία σε αυτό. Έχω μία ερώτηση κάθε κράτος μέλος έχει μία στατιστική αρχή. Εσείς απευθύνεστε λοιπόν στις εθνικές στατιστικές αρχές, είπατε, όχι μόνο στη Eurostat. Η ερώτηση μου είναι, υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη στατιστική αρχή. Ένα. Δύο. Σας δίνω στοιχεία για τις υπηρεσίες. Έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες της. Κατόπιν, σωστά αναφερθήκατε στη σχέση που υπάρχει μεταξύ αγαθών, υπερ, ε, υπηρεσιών, ίντερνετ των πραγμάτων, ε, ρομποτική, αυτοματοποίηση κλπ. Υπάρχει δυνατότητα να διακρίνετε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή μπορείτε να διακρίνετε υπηρεσίες από, αγαθές, από αγαθά ή εμπορεύματα ή δεν μπορείτε να κάνετε διάκριση μεταξύ των συμβάσεων. Γιατί αυτό θα ήταν καλό να το δούμε. Τώρα, οι διαγωνισμοί, οι κρατικοί διαγωνισμοί. Μιλήσατε για χώρες που θέλατε να καλύψετε. Η ερώτησή μου είναι, έχετε κάνει σύνδεση μόνο με τα κράτη ή και με υποκείμενες δομές, περιφέρειες, επαρχίες κλπ. Αν θυμάμαι καλά, για την Ιαπωνία είχαμε φτάσει μέχρι το επίπεδο των Δήμων. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τα στοιχεία που έχετε είναι μόνο σε επίπεδο κράτους ή και σε χαμηλότερα επίπεδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Μία ερώτηση για τις στατιστικές, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως. Χαίρομαι που έχουμε ένα κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις συμφωνίες ελευθερών εμπορίου της νέας κοπής. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο δυναμικό για εμπόριο. Για τις στατιστικές λοιπόν που έχετε μέχρι στιγμής μπορεί να φτάσετε σε κάποια πορίσματα χάρη σε αυτές τις στατιστικές που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε και να βελτιώσετε τα κεφάλαια για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, ούτω ώστε να έχουμε περισσότερες πολιτικές που διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έφτασα εγκαίρως, ήμουν σε μια άλλη επιτροπή και θέλω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Όλη αυτή η πληροφορία είναι σημαντική για να αυξηθεί η διαφάνεια, που είναι σημαντικό στοιχείο για να διευκολύνουμε ε, την ισοτιμία στο πεδίο αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε το εξή. Όταν πάμε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία μια τρίτη χώρα, ειδικά οι συμφωνίες που έχουν τις ε, δημόσιες προμήθειες. Γιατί δεν απαιτούμε να σέβονται τους κανόνες του ΠΟΕ σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Γιατί υπάρχουν τέτοιες χώρες που ξεχνούν σε ό,τι αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, τους κανόνες του ΠΟΕ για το πεδίο αυτό. Δεν θα πρέπει να τις καταστήσουμε προϋπόθεση στις ε, συμφωνίες αυτές. Το να σέβονται τους κανόνες ΠΟΕ οι χώρες αυτές. Πώς θα σέβονται τους κανόνες σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες, πώς θα παίζουν με βάση τους κανόνες οι τρίτες χώρες. Δύο ερωτήσεις και από πλευρά μου, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτον, για την σημασία των ε, υπηρεσιών. Έχουμε πολλές εμπορικές συμφωνίες με τις αφρικανικές χώρες ειδικά, όπου υπάρχει δυνατότητα για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν εδώ, στην Ευρώπη. Ίσως οι αφρικανικές χώρες θα... Καλό θα ήταν να εστιάσουν στην, ε, στις υπηρεσίες παρά στην ε, παραγωγή αγαθών τύπου μηχανήματα ας πούμε. Γιατί δεν θα ήταν τόσο ανταγωνιστικές. Έχετε στοιχεία από την ε, εισαγωγή υπηρεσιών που έρχονται από αφρικανικές, προέρχονται από αφρικανικές χώρες. Και δεύτερον, για τις κρατικές προμήθειες. Έχουμε νέα νομοθεσία για τα IPI, για τις συμφωνίες αυτές ελευθέρου εμπορίου. Αναφέρατε την ε, Ιαπωνία, την Κίνα, τους βασικούς μας εταίρους. Έχουν την τάση να κλείνουν τις αγορές τους ή είναι Ανοιχτέ οι χώρε αυτές. Πολύ σημαντικές, πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσεις. Θα απαντήσω με τη σειρά που τις άκουσα για τη συμμετοχή των κρατών μελών και τα διαθέσιμα στοιχεία. Η Eurostat έκανε τεράστια προσπάθεια για να ετοιμάσει τόσο λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες για όλα τα κράτη-μέλη και για εκείνα ακόμα που δεν συμμετέχουν στο εγχείρημα. Υπάρχει μια μεθοδολογία του ΟΗΕ που εφάρμοσε η Eurostat με τη βοήθεια των λίγων χωρών που μπήκαν σε αυτό το project και λίγο-λίγο φτιάξαμε μια αξιόπιστη βάση δεδομένων, ακόμα και για χώρες με πληροφορίες, δηλαδή και για χώρες που δεν συμμετείχαν στο project αυτό δίνανε εξηγήσει στα δεδομένα, αλλά δεν υπέβαλαν τα δεδομένα τους. Καλό θα ήταν να πείσετε αυτές τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, που καμιά φορά δεν είναι μικρές χώρες, έτσι. Είναι μεγάλες και αξιοσέβαστες στατιστικές υπηρεσίες που έχουν τους δικούς τους λόγους και δεν θέλουν να παίξουν ενεργό ρόλο. Αν μπορείτε να τους, να τους ε, πείσετε ε, να συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα. Έχουμε λοιπόν πολύ καλή βάση δεδομένων αλλά για να βελτιωθεί θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν πιο ενεργά. Η κατάσταση τώρα είναι πιο δύσκολη για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες από αυτές, γιατί δεν υπάρχει μεθοδολογία του ΟΗΕ που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Eurostat και το να χρησιμοποιεί τις ε, πληροφορίες που έχουν εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και από αυτές να κάνει κάποιες εκτιμήσεις είναι δύσκολο. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε στοιχεία ε, μόνο από τα κράτη-μέλη που αποφασίζουν να υποβάλουν τα δεδομένα τους. Χωρίς τη συνεργασία του κράτους μέλους τίποτα δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία για τις μικρομεσαίες. Και στηρίζω τη δήλωσή σα ότι οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις είναι πολύ πιο σημαντικές από ό,τι νομίζαμε. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο για αυτέ είναι και η απόδειξη αυτού του γεγονότος. Ε, αλλά συνολικά όλα τα κεφάλαια των συμφωνιών ελεύθερων μπορεί να βοηθήσουν μέσα σε όχι μόνο το ειδικό κεφάλαιο για αυτέ. Ε, λοιπόν Έχουμε κάνει πολλαπλέ προσπάθειε για να καταλάβουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και τα εμπόδια που αντιμετωπίσουν. Πριν από κάνα δύο χρόνια είχαμε ένα project για τι μη δασμολογικέ τροχοπέδε που ε, αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίε. Ε, για του κανόνε καταγωγή, α πούμε, και σε ποιο βαθμό μπορούν να του σεβαστούν οι επιχειρήσει αυτέ. Ε, Επίση για τι υπηρεσίε. Ρωτάμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει τι μεταβλητές αντιμετωπίζετε για να μπορέσετε να δώσετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, αν τα βάλουμε, βάλουμε όλες αυτές τις ψηφίδες, θα φτιάξουμε καλύτερη εικόνα. Και αν χρειαστεί να αλλάξουμε και τους σημερινούς μας κανόνες. Ε, πιστεύουμε ότι οι κανόνες, έτσι πιστεύουμε ότι οι κανόνες μας είναι καλοί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αλλά είμαστε ήδη σε καλή βάση για τις δημόσιες προμήθειες, κρατικές προμήθειες και τα δεδομένα και το επίπεδο ανάλυσης. Στις χώρες που ανέφερα στη διαφάνεια, σε όλες αυτές τις χώρες σχεδόν, έχουμε την τύχη να έχουμε δεδομένα πέρα από το εθνικό επίπεδο. Έχουμε, ας πούμε, δεδομένα για τους Δήμους και τις κοινότητες στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Βραζιλία. Αλλά συλλέγουμε δεδομένα για τις, ε, συμβάσεις που σέβονται τα διεθνή πρότυπα. Δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα για τις συμβάσεις, ας πούμε, 50.000 ευρώ χαμηλή αξία, ας πούμε. Δεν έχουμε διεθνείς κανόνες, ας πούμε, για να εμποδίσουμε τις διακρίσεις σε αυτά τα μικρά συμβόλαια. Αν όμως η σύμβαση είναι πάνω από ένα κατόφλι και εκεί υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις, Νομίζω 130.000 ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα έχουμε κανόνες που τους έχουμε διαπραγματευτεί στις συμφωνίες ε, ελευθερών εμπορίου με τον ΠΟΕ. Εκεί εστιάζουμε. Αν θέλουμε και άλλες πληροφορίες, ε, αν έχουμε και άλλες πληροφορίες, τις συλλέγουμε δηλαδή. Ακόμα και για πιο μικρές συμβάσεις. Αλλά γενικά μπορώ να σας πω ότι ξεπερνάμε το κεντρικό εθνικό δηλαδή επίπεδο. Έχουμε πλήρη δεδομένα ακόμα και για δήμους και κοινότητες από αυτές τις χώρες που σας ανέφερα στη διαφάνεια για τις προμήθειες. Ίσως θα πρέπει να ομαδοποιήσω και να απαντήσω συνολικά σε αυτές τις ερωτήσεις πριν πάω στην, ε, στις υπηρεσίες και στην Αφρική. Αυτά τα δεδομένα θα ήταν σημαντικά, όχι μόνο για τις συμφωνίες ελευθερών εμπορίου και για τις διαπραγματεύσεις μας, αλλά και στις διμερείς συζητήσεις ε, και τις πρωτοβουλίες που έχουμε για το, τις προμήθειες, για να καταλάβουμε πώς η πρόσβαση στην αγορά ε, λειτουργεί και αν οι εταιρείε μας αντιμετωπίζονται ισότιμα στις τρίτες χώρες. Υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Καταρχάς, ε, πληροφορίε ε, για τι συμβάσει παλιά δεν είχαμε, τώρα τι έχουμε. Έχουμε πλήρη ταξινόμηση που βασίζεται σε μια ταξινόμηση ε, εγκεκριμένη ε, από τον ΟΣΑ. Μια χώρα που λέει δεν θα κερδίσει μια ευρωπαϊκή εταιρεία τη σύμβαση, το λαμβάνουμε υπόψη. βλέπουμε τι διακρίσεις υπάρχουν τι διαδικαστικά εμπόδια υπάρχουν με την δυνατότητα που έχουμε να κερδίσουμε συμβάσεις. Ε, ακόμα δεν έχουμε πλήρως τα δεδομένα. Ε, όλο και περισσότερο έρχονται δεδομένα και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα τα αναλύσουμε για, τα, για αυτά τα 38 εκατομμύρια συμβάσεις για να καταλάβουμε τα προβλήματα, για να επιταχύνουμε τις προσπάθειες εφαρμογής μαζί με το βασικό αξιωματούχο για, υπεύθυνο για θέματα εφαρμογής των συμφωνιών. Τώρα, ILO και άλλες ε, προϋποθέσεις μπορούμε να τις συνδέσουμε και αυτές με τις προμήθειες. Τα δεδομένα μας δεν φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας. Δεν έχουμε δεδομένα για το αν η χώρα σέβεται κάποια πράγματα, αν έχει εφαρμόσει και σεβαστεί οι συμβάσεις του ILO. Γιατί αν υπήρχαν, ε, ούτως ή άλλως θα, εφαρμοζόταν συλλογικά για όλες τις συμβάσεις. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να επαληθεύσει αυτές τις α, ε, πληροφορίες, ε, τις λεπτομέρειες πληροφορίες, με τις γενικές πληροφορίες που έχουμε για τη συμμόρφωση της χώρας με τους κανόνες. Δεν το κάναμε όμως κατά ανάγκη. Όμω, ε, έλειπε αυτό το κομμάτι. Τώρα η υπηρεσία στην Αφρική, έχουμε κάποιες πληροφορίε για τις εισαγωγέ. Να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό που σας έδειξα για τις εξαγωγέ ε, το έχουμε και για τις ευρωπαϊκές εισαγωγέ με ίδιε λεπτομέρειες. Για το αφρικανικό εμπόριο ε, βασιζόμαστε στις στατιστικέ ε, πληροφορίε και την ποιότητά του ε, που μα δίνουν αφρικανικέ χώρε. Και δεν είναι ακριβώ το ίδιο επίπεδο όλε. Κάποιε βασικέ αφρικανικέ χώρε έχουν σχετικά καλά δεδομένα που καταλαβα... μα δίνουν μια εικόνα αρκετά καλή για το είδο του εμπορίου που κάνουν στι ε, υπηρεσίε, ε, ενώ ορισμένε χώρε δεν έχουν καμία πληροφορία. Δεν μα δίνουν καμία πληροφορία. Αυτό που βλέπουμε ότι για μια αφρικανική χώρα που ενδιαφέρεται στην προώθηση του εμπορίου στις ε, υπηρεσίες, ε, όπως η Κένια ας πούμε, ε, η οποία μοιάζει με την Ινδία, εκεί έχουμε πολλές πληροφορίες. Βασίζεται η Κένια στις ψηφιακές υπηρεσίες. Το ΜΟΤ είναι πολύ σημαντικό, εργατικό, δυναμικό. Βεβαίως δεν έχουν την ίδια δυνατότητα να επενδύσουν όπως η Ευρώπη. για την εξαγωγή άλλων υπηρεσιών ε, πέρα του τουρισμού, η λύση ε, είναι στην ψηφιακή οικονομία. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που έχουμε μια βάση δεδομένων. Γιατί συχνά οι συζητήσεις μας, παρότι η Επιτροπή είναι θαυμάσια βέβαια, ε, δεν γίνεται βάση στοιχείων. Οπότε είναι χρήσιμο να έχουμε στοιχεία πια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ένα σχόλιο που αφορούσε την τελευταία διαφάνεια. Ο πρώτος μου, το πρώτο μου αφεντικό στον ΟΗΕ είπε ότι χωρίς καλά δεδομένα προχωράμε στα τυφλά. Και αν δεν βλέπεις ποιο είναι το πρόβλημα, πώς θα το διορθώσεις. Εμείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε ακριβώς αυτό να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε τα δεδομένα για να μας καθοδηγήσουν. Μερικές φορές χρειαζόμαστε, πρέπει να περάσουν 25 χρόνια για να συλλέξουμε καλά δεδομένα, αλλά δεν σταματάμε, είμαστε άοκνοι μέχρι να τα συλλέξουμε. Πολύ ωραία. Κλείσαμε το σημείο 10 και πάμε στο 11. Το αγαπημένο μου. Τα διάφορα. Τίποτα. 12. Η επόμενη συνεδρίαση, συνεδριάσεις, Δευτέρα, στις 30 έχουμε την ακρόαση του Φιλ Χόγκαν καταρχήν. 30 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα. Και η επόμενη τακτική συνεδρίαση θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου, 9 η ώρα. Τελειώσαμε. Καλή εβδομάδα.